Συνάδελφοι, να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Σημείο υπαριθμών 13. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Ρωμάνα Βλαχούτιν, πρέσβυρα με ειδική αποστολή για τη συνδεσιμότητα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τον Προντάν. Πολλές φορές την είχαμε εδώ στην Επιτροπή μας, ε, την κυρία Βλαχούτιν ως ειδική απεσταλμένη στα τύρανα, αλλά τώρα έχει έναν τελείως διαφορετικό ρόλο πλέον. Η πρόσκληση που σας απευθύναμε αποτελεί και μια συνέχεια της πρωτοβουλίας του συναδέλφου μας Reinhard Bütikofer που ζήτησε να συζητηθεί το θέμα της συνδεσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ημερησία διάταξη. Είναι ένα θέμα που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία και όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις, την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή έχουμε καθυστερήσει λίγο, ίσως θα μπορούσατε να κάνετε μια μικρή εισήγηση, δεκάλεπτη θα έλεγα, και από εκεί και πέρα θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε θέματα μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ, είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Η συνδεσιμότητα είναι ένα πολύ ευρύ θέμα. Οπότε θα ήθελα να χωρίσω την εισήγησή μου σε δύο τμήματα. Πρώτον, να μιλήσω γενικά για τη συνδεσιμότητα και τι, ποια είναι η σημασία για την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια, τις οικονομίες μας και από εκεί και πέρα θα μπω και σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διασύνδεση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασίας και τι έχουμε κάνει στον τομέα αυτό μέχρι στιγμής. Με ρωτούν πάντοτε τι είναι η συνδεσιμότητα και τι σημαίνει ο όρος αυτός. Γιατί φυσικά διάφορα ακροατήρια ε, την ερμηνεύουν την έννοια με διαφορετικό τρόπο. Στην ουσία, αν υπάρχουν πολλές απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα, είναι μια ολοκληρωμένη επένδυση σε επενδύσεις, ε, σε μια, μια ολοκληρωμένη επένδυση σε υποδομές και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε, είναι η ίδια ένα αποτέλεσμα συνοχής και ολοκληρωμένων επενδύσεων. Γιατί έχουμε γίνει αυτό που έχουμε γίνει ακριβώς επειδή έγιναν σχετικές ολοκληρωμένες επενδύσεις σε υποδομές. Και ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η συνδεσιμότητα δεν είναι ουδέτερη όσον αφορά την αξία της συνοδεύεται από κανονισμούς, από κανόνες, από ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος, ισότητα φύλων, κοινωνικά δικαιώματα και ευρωπαϊκό όραμα ως προς την παγκόσμια διακυβέρνηση. Θέλω να διατρέξω μαζί σας ε, δύο-τρία βασικά στοιχεία και επιπτώσεις της συνδεσιμότητας στην εξωτερική πολιτική μας. Πρώτον, υπάρχει μια πολιτική επίπτωση. Αν δείτε τους αριθμούς και έχουμε κάνει πολλές έρευνες, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται πάνω-πάνω στους περισσότερους πίνακες κατάταξης ε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε μεγάλο ΑΕΠ, εμπορικές συναλλαγές, έχουμε μεγάλο ποσοστό επενδύσεων, περισσοκών στοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ε, ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο. Όμως υπάρχει μια ενδιαφέρουσα σύγκριση. Στον τελευταίο δημοσιονομικό κύκλο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της παρήχαν 414 εκατομμύρια ε, ευρώ ε, σε επιδοτήσεις ε, σε σύγκριση με τα 400 δις που έγιναν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Belt and Road. Όμως η, η, η απήχηση είναι διαφορετική, γιατί τα ίδια χρήματα δεν μετα, μετουσιώνονται πάντοτε στην ίδια πολιτική, αν θέλετε, στον πολιτικό αντίκτυπο. Η Ευρώπη πρέπει από δωρητής ή τέλος πάντων πάροχος να γίνει ένας πραγματικός παίκτη για να αποκτήσει την πραγματική ουσία της ε, ικανότητάς της να παρεμβαίνει. Όλα αυτά βεβαίως σχετίζονται και με την οικονομική μας ανάπτυξη, με τη συνοχή μας, θα υπησέλθω σε αυτά αργότερα. Ιδίω ε, στη συνέχεια μάλλον, όσον αφορά, είναι πάρα πολύ σημαντική η συνδεσιμότητα για την οικονομική ανεξαρτησία και ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διπλή χρήση εγκαταστάσεων όπως οι λιμένες, πρόσβαση σε πρώτες ύλες, η συζήτηση για το 5G, αλυσίδες αξίες. Και νομίζω και η τελευταία κατάσταση με τον κορονοϊρό και την, ε, την ε, διατάραξη των προμηθειών είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα γιατί υπάρχουν σαφείς αναφορές ότι αν δεν εξομαλυνθεί σύντομα η κατάσταση ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε σημαντική έλλειψη φαρμακευτικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων και αντιβιωτικών. Γιατί το 77% των γενώσιμων φαρμάκων παράγονται στην Ινδία και άρα και εκείνοι εξαρτώνται με τη σειρά τους από τις εισαγωγές από την Κίνα. Και ένα επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο για μας είναι η οικονομική ευημερία και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η ε, έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας κατέδειξε ότι κάθε ποσοστο, ποσοστιαία μονάδα που επενδύεται σε υποδομές ε, οδηγεί σε ανάπτυξη 2% και σε αναπτυσσόμενες χώρες 7%. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό σημαίνει και μεγαλύτερη πρόσβαση σε αγορές και ανάπτυξη ε, σε ε, ε ύψους 1 έως 1,5% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 4-4,5% στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα χρήματα, είναι, το κεφάλ, τα, τα κεφάλαια είναι σχετικά φθηνά αυτή τη στιγμή και στην ευρωπαϊκή κεφαλαία αγορά υπάρχει ένα τρισεκατομμύριο διαθέσιμο για επενδύσεις. Ταυτόχρονα υπάρχουν τεράστιες ανάγκες. Υπάρχουν προβλέψεις ότι μόνο στην Ασία έως το 2030 θα πρέπει να επενδυθούν γύρω στα 36 τρισεκατομμύρια ευρώ και αυτά δεν μπορούν να εξευρεθούν μόνο από κρατικά ταμεία. Οπότε πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να γίνουν ιδιωτικέ επενδύσει και ιδιωτικοί Ευρωπαίοι φορεί να συνεργαστούν μαζί μα για το θέμα τη συνδεσιμότητα σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλοι λοιπόν μιλούν για τη συνδεσιμότητα γιατί πραγματικά έχει καταστεί ένα γεωπολιτικό εργαλείο στον αιώνα μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως ανταποκρίνεται στην πρόκληση αυτή. Τον Οκτώβριο του 2018 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το τη στρατηγική για τη διασύνδεση Ευρωπαϊκής Ένωση Ασία και, το, και στις αρχές του 2019 ξεκίνησε η υλοποίηση. Αρχικώ κάνοντας μια εσωτερική οργάνωση, δηλαδή στην ΕΕΔ, δημιουργήθηκε η θέση του πρέσβη με ειδική αποστολή για τη συνδεσιμότητα, υπάρχει μια μικρή ομάδα, υπάρχει μια ιδιοπηρεσιακή ομάδα όπου ε, συμπροεδρεύουμε με συναδέλφους από την Κομισιόν και στην ουσία συντονίζουμε όλη αυτή τη διαδικασία και με εκπροσώπους των κρατών μελών. Η ίδια η στρατηγική κατοχυρώνει βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής προσέγγισης. Υπάρχουν τέσσερις πυλώνες που χρησιμοποιούμε, μεταφορές, ενέργεια, ψηφιοποίηση και ανθρώπινη συνδεσιμότητα. Έργα ε, που θέλουμε να, να ολοκληρώσουμε είναι η κατασκευή φυσικών εγκαταστάσεων, η εξασφάλιση χρηματοδοτικής στήριξης και η δημιουργία εταιρικών σχέσεων με ε, χώρες και περιοχές που σκέφτονται με παρόμοιο τρόπο. Και υπάρχουν και, και οι στόχοι που είναι η βιωσιμότητα, ε, η περιβαλλοντική, κοινωνική βιωσιμότητα και η όρια ανταγωνισμού. Επίσης έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις με πιθανές χώρες δικαιούχους καθώς και κοινότητες επιχειρηματιών καθώς και εκείνους που ερευνούν το ζήτημα της ε, συνδεσιμότητας, γιατί θέλουμε πάντοτε να βασίζουμε το σχεδιασμό μας σε επιστημονικές ενδείξεις και στοιχεία. Στο μεσοδιάστημα διαπραγματευτήκαμε και μια εταιρική σχέση συνδεσιμότητας με την Ιαπωνία και το Σεπτέμβριο πέρσι έγινε και ένα εξαιρετικά επιτυχημένο φόρουμ για τη συνδεσιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που οδήγησε στην αλληλεπίδραση με 11,5 εκατομμύρια πολίτες μέσω των ε, social media. Οι εργασίες σχετικά με την υλοποίηση επίσης έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα ως προς το που υπάρχουν ελλείψεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ποια είναι τα, τα πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια είναι η δυναμική, ποιες αποφάσεις πρέπει να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να ηγηθεί στον τομέα τη συνδεσιμότητας και πέραν των συνόρων της. Για τι ελλείψει, ένα από τα βασικά προβλήματά μας είναι ο εκτεταμένος κατακαιρματισμός. Πολλά κάνουμε, κάνουμε πολλά, αλλά Υπάρχουν πάρα πολλά ιδρύματα, χώρε, ε, υπηρεσίε, με διάφορα κτικόληξα, διάφορα ονόματα, διάφορου τίτλου, διάφορου νομικέ προσωπικότητε και πολλέ φορέ δεν είναι εύκολο να διαμορφώσει μια συνολική εικόνα για το τι γίνεται. Και αυτό δεν είναι μόνο επικοινωνιακό πρόβλημα. Δεν είναι ότι δεν ξέρουμε πώ ακριβώ να επικοινωνούμε μεταξύ μα. Είναι και ένα συστημικό ζήτημα, διότι πηγάζει από διάφορα παράλληλα στοιχεία ή επίπεδα δράση. άρα πρέπει και εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτό και μέσω των νέων εργαλείων και μηχανισμών προγραμματισμού και σε συνεργασία με την ε, Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται προφανώς μια συνολική συστημική προσέγγιση, ενιαία και ομοιόμορφη και βεβαίως τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να έχουν μια παγκόσμια παρουσία μόνο ενωμένα. Δεν μπορεί ούτε το κάθε κράτος ξεχωριστά ούτε κάθε ένα θεσμικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο του. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Το ΠΔΠ προβλέπει αρκετά χρήματα, σημαντικά χρήματα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιωσιμότητας ΣΥΝ που είναι και εκεί ένας, ένας μηχανισμός που μπορεί να, να προωθηθεί η συνδεσιμότητα. Επίσης, έχουμε έλλειψη μιας ενιαίας πλατφόρμας χρηματοδότησης, ένα, ενός μηχανισμού όπου δηλαδή δημόσιες και ιδιωτικές, δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν για επενδύσεις. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αν είχαμε ένα τέτοιον μηχανισμό εξορισμού θα μας ε, οδηγούσε σε πολύ μεγαλύτερη συνεκτικότητα και συνοχή ως προς το τι κάνουμε στον τομέα της συνδεσιμότητας. Και τέλος πρέπει να αναδείξουμε μια ρητή, απερίφραστη ε, φιλοδοξία η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει έναν γεωπολιτικό ρόλο, να αποτελέσει έναν αξιόπιστο εταίρο στον τομέα της συνδεσιμότητας με βάση τη δική μας ευρωπαϊκή αντίληψη, βεβαίως και για τους ίσους όρους ανταγωνισμού. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο αυτό. Μας δίνει μια τέτοια στρατηγική τη δυνατότητα να σημειώσουμε πρόοδο και συζητήσεις με, τον, με τους εταίρους μας. Η ευρωπαϊκή στάση λοιπόν πρέπει να είναι συνεκτική, συνολική, φιλική στον ε, ε χρήστη. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια ώστε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τα... Ας ακούσουμε τώρα τους συναδέλφους που θα ήθελαν να συμμετάσχουν στην συζήτηση αυτή. Αναφερθήκατε στη δυνατότητα, την αστήρευτη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργεί ακρόνημα. Εγώ είμαι εδώ και χρόνια φαν τουλάχιστον ετησίας απαγόρευσης νέων τέτοιων ακρονίμων. Έχουμε ένα σωρό αστεία παραδείγματα. Το «Εντίτσι» είναι το τελευταίο παράδειγμα, δεν ξέρουμε καν πώς να το προφέρουμε. NDICI, NDICI, ό,τι θέλετε. Κανείς εκτός του Μπερλεμό ή της έδρας της ΕΙΕΔ δεν θα έχει ιδέα πώς να τα προφέρει όλα αυτά. Δεν πειράζει. Ας ακούσουμε τώρα τους ε, συναδέλφους, ε, τον συνάδελφο που το έθεσε το θέμα αυτό, ο κύριος Μπιουτικόφα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Βλαχούτιν για την παρουσίαση αυτή. Χαίρομαι που το εξετάζουμε αυτό το θέμα στην ΑΦΕΤ γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι η ίδια μας η φιλοδοξία η γεωπολιτική που φαντάζομαι να την συμμερίζεται και η Επιτροπή λέει ο Μιλτής ορίζει ότι η πολιτική της πληροφορίας και της συνδεσιμότητας θα ήταν ένα από τα πιο σημαντικά μέσα και μάλλον θα πρέπει να μας ενθαρρύνει αυτό να προωθήσουμε το θεματολόγιο αυτό που βλέπουμε ότι άλλοι τον παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον. Οι Αμερικανοί, επί παραδείγματι, έχουν κάτι περισσότερο από ενδιαφέρον να συνεργαστούν μαζί μας μέσω διαφόρων μηχανισμών μέσω του δικού τους ε, δικτύου Blue Dot Η κυρία Βλαχούτιν ήδη μας ανέφερε για την Ιαπωνία που υπέγραψε συμφωνία. ότι ω Κορέα είναι απολύτως πρόθυμη και ακούω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από τις χώρες Ασιαν. Επομένως, όλα αυτά αποτυπώνουν μια προσδοκία πρώτων πυλών στο κατόφλι μας, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να εκπληρώσουμε τις ε, υποσχέσεις μας, υλοποιώντας όλη αυτή την συνδεσιμότητα. Θυμάμαι και μια πολύ πρόσφατη συζήτηση με τον Υπουργό Οικονομικών της Ινδονησίας και όταν ερωτήθηκε η κυρία Υπουργός τι πιστεύει για την ε, στρατηγική της Κίνας, το Belt and Road, απήντησε ότι δώστε μου μια εναλλακτική και θα σας πω τι πιστεύω. Και είναι ενδιαφέρον γιατί ε, όχι μόνο για χώρες σαν την Ινδονησία, δηλαδή εάν αυτή τη στρατηγική της συνδεσιμότητας μπορούμε να, τη, δώσουμε πνοή, φτερά, ρόδες θα έχουμε πολύ, μια πολύ καλή ευκαιρία συνεργασίας όχι μόνο προς την κατεύθυνση της Ανατολικής Ασίας αλλά και προς την Αφρική. Τώρα υπάρχουν ένα-δύο θέματα προτεραιότητας που πρέπει να δούμε αν θέλουμε να πετάξει αυτή η στρατηγική, δηλαδή να ακολουθήσουμε τις υποσχέσεις μας από κάποια χρηματοδότηση, κονδύλια, όπως είπατε και το Ιντίτσι, εκεί παίζεται το παιχνίδι. Το οποίο δεν σημαίνει απλώς να και τοποθετήσουμε τα κατάλληλα κονδύλια πίσω από την χ γραμμή του προϋπολογισμού, θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε ένα μέσο που έχει υλοποιηθεί σε κάποιες περιφερειές αλλά όχι στην Ασία. Θα ήταν καλό να επεκταθεί ώστε να συμπεριλαμβάνει και τις ασιατικές χώρες. Και θα υπέθετα επίσης ότι καλό θα ήταν να ενθαρρύνουμε, να υποστηρίξουμε και την Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα για τα Δεραθρωτικά να γίνουν πιο σημαντικοί παίκτες. Και πέραν των όσων κάνει η ομάδα συνδεσιμότητας, χρειαζόμαστε πιο εμφανή υποστήριξη από τα υψηλότερα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή είτε η ίδια η Πρόεδρος θα πρέπει να τα αναλάβει είτε ένας από τους εκτελεστικούς αντιπροέδρους να καταστεί τσάρος του θέματος και να αναλάβει το θεματολόγιο αυτό που είναι ευρύτατο. Γιατί υπάρχει και προφανής και αόρατη αντιπολίτευση έναντι του γεωπολιτικού αυτού προγράμματος. Απαιτείται μια συντονισμένη προσπάθεια από την κορυφή για να τροχοδρομήσει αυτό το όραμα. Και θα αντιφάσκαμε αν δεν το βοηθούσαμε. Πόσο μάλλον που είδαμε και το μεγάλο ενδιαφέρον μετά την εκδήλωση του περασμένου Σεπτεμβρίου που μπορεί να εξανεμιστεί βεβαίω. Αν για μία ακόμα φορά δοθεί το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε διάφορα ωραία πράγματα αλλά δεν τα παρακολούθησε με πράξεις, θα είναι άλλη μια χαμένη ευκαιρία. Ελπίζω πραγματικά να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ώστε να μην είναι έτσι τα πράγματα. Ευχαριστώ κυρία Μπιουτικόφα, η κυρία Φωτίγκα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ τον κύριο Πρέσβη για την εισήγησή του. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπιουτουικόφα για την πρωτοβουλία. Υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές του θέματος αυτού που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής πέραν των υφισταμένων πολιτικών μας. Η σημασία του ζητήματος αυτού είχε δοκιμαστεί όχι πολλά χρόνια πίσω, πριν από δύο νομίζω χρόνια. Είχα ταξιδέψει από το Ελσίνκι στη Σόφια με αεροπλάνο και αυτό μου πήρε όλη την ημέρα, χωρίς να υπάρχουν καθυστερήσεις, λέει η κυρία Φωτίγκα. Ήταν εντυπωσιακό. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι πρέπει να δούμε τις ανταποκρίσεις μας, τις συνδέσεις μας και εντός και εκτός της Υπήρου θα ήθελα να αναφέρω δύο στοιχεία. Οι θαλάσσιες συνδέσεις με την Ιαπωνία έχουμε την ανάγκη να εξασφαλίσουμε την ελευθερία της ναυσιπλοείας που είναι και το χόμπι μου λέει η κυρία Φωτίγκα και πρέπει πολύ γρήγορα να υιοθετήσουμε και μια αφρικανική στρατηγική. Από ό,τι ακούω αυτή είναι η πρόθεση για τις αρχές του Μαρτίου ώστε να εστιαστούμε και σε αυτό γιατί πρέπει να μην ξεχνούμε ότι οι μεταφορές και οι υποδομές εκεί είναι ακόμα πολύ πρώιμες. Και είναι και η δυνατότητα σύνδεσής μας με τις πρωτεύουσες παρακτήων χωρών χωρίς να μπορούμε να βοηθήσουμε καθόλου την ενσωμάτωση των αφρικανικών αγορών ό,τι και να πιστεύουμε για την περιφερειοποίηση ή το G5 ή τις ανατολικές αφρικανικές χώρες υπάρχει το τεράστιο εμπόδιο των μεταφορών και της συνδεσιμότητας. Thank Further comments from yours. Ευχαριστώ την κυρία Φωτίγκα. Δεν βλέπω να έχουμε άλλα σχόλια. Εκτός μικροφώνου. Μικρόφωνο. Sorry, sorry. Ε, κύριε Μπουτικόφερ, ε, είπατε δώστε μου μια εναλλακτική λύση. Είναι μια πρόταση που την ακούμε πολύ συχνά με τους συνομιλητές μας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είχα παρόμοιες συζητήσεις στην Κεντρική Ασία, γιατί αυτή η στρατηγική καλύπτει ε, περιοχές από την Ευρώπη μέχρι την Ασία, καλύπτει τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ανατολική Γειτονία, την Κεντρική Ασία και την ίδια την Ασία. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας να δημιουργήσουμε μια εναλλακτική που να μην είναι μόνο στιβαρή από πλευράς ε, οικονομικής προσφοράς, αλλά που να εστιάζεται, που να είναι επικεντρωμένη και κατανοητή. Η συνδεσιμότητα απαιτεί ε, κλίμακα και για να έχεις ουσιώδεις αλλαγές θα πρέπει να το κάνεις σε μια κλίμακα που να επιφέρονται αυτές οι αλλαγές. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σε περιφερειακό επίπεδο επίσης. Αναφερθήκατε επίσης και σε άλλους εταίρους, άλλες ε, δυνατότητες. Πρέπει να σας πω ότι η Ινδία ενδιαφέρεται πάρα πολύ στο, σε μεγαλύτερη συνδεσιμότητα με εμά, η Ινδία είναι μια συναρπαστική ευκαιρία. Είναι κάτι που σίγουρα θα παρακολουθήσουμε. Η περιοχή των χωρών ΑΣΕΑΝ επίσης αποτελούν μεγάλη ευκαιρία για αρκετές από τις επιχειρήσεις μα που δραστηριοποιούνται εκεί. Αλλά αυτό που είναι κλειδί στο να γίνει αυτό με συνεκτικό τρόπο είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο και τα πρότυπα που συνοδεύουν τις επενδύσεις και τις υποδομές, διότι αυτό μας καθιστά ανταγωνιστικούς ή καθιστά τις επιχειρήσεις μας ανταγωνιστικές. Και είναι προς το συμφέρον μας να στηρίξουμε το επίπεδο των ε, προτύπων που κατά την άποψή μας είναι προς όφελος της βιωσιμότητας αυτών των έργων μα μας έχουν προσεγγίσει οι ΙΠΑ για να ε, δούμε το δίκτυο Blue Dot και την ιδέα της πιστοποίησης των υποδομών καλής ποιότητας. Επίσης, συνεργαζόμαστε με την Ιαπωνία στην υλοποίηση της ε, συμφωνίας. Αυτό που είναι καινοτόμο στη δουλειά με την Ιαπωνία είναι ότι έχουμε εντοπίσει πέντε περιφέρειες όπου θέλουμε να συνεργαστούμε. Έχουμε Δυτικά Βαλκάνια, Ανατολική ε, περιοχή, Αφρική, Ανατολική Ασία, και Ανδρική Ασία και αυτό που θέλω να τονίσω είναι σημαντικό για μας να δώσουμε κίνητρα στην ιδιωτική επένδυση. Αυτό απαιτεί, προϋποθέτει ιδιωτικά κεφάλαια, ειδικού ε, ιδιωτικές επιχειρήσεις και έχουμε συνεργαστεί με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και πρέπει να πω κατανοούν πλήρως αυτό που διακυβεύεται. Υπάρχει ένας αριθμός επιχειρήσεων από την Ιαπωνία, 69% γερμανικών επιχειρήσεων πάνε στην Ιαπωνία, όχι για την Ιαπωνική αγορά, για να, για να συνεργαστούν με Ιαπωνικές ε, επιχειρήσεις, για να σχηματίσουν κοινοπραξίες εκεί. Και αυτό είναι ένα καλό μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να ακολουθηθεί και σε άλλους τομείς επίσης. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν οποιαδήποτε περαιτέρω σχόλια. Δεν ε, βλέπω να ισχύει αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε κυρία Πρέσβης και θα παρακολουθήσουμε αυτό το θέμα της συνδεσιμότητας και είναι καλή αυτή η πρώτη ενημέρωση των δραστηριοτήτων σας. Ε, συνάδελφοι, το επόμενο σημείο προβλέπεται για τις 5 παρατέταρτο. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτών. Στις 5 παρατέταρτο θα... Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε εδώ μαζί αρκετούς Ισπανούς συναδέλφους για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Καλό απόγευμα σε όλους. Buenas tardes, λέει ο Πρόεδρος. Να συνεχίσουμε. Το τελευταίο σημείο στην ε, διάταξή μας είναι ανταλλαγή απόψεων ενημέρωση από την ΕΕ για την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Η κυρία Βερονίκ Λορένσο, επικεφαλής του τμήματος Νότια Αμερική της ΙΕΒ. Μετά ένα χρόνο αργότερα από την εκλογή του κυρίου Γκουαϊντό Προέδρου της ε, η κατάσταση δεν έχει αποκλιμακωθεί κάθε άλλο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει και υποστηρίζει τον Χουάν Γκουαϊντό ως πρόεδρο του Κοινοβουλίου και ως νόμιμο εκπρόσωπο υπό το Σύνταγμα της Βενεζουέλα μεταβατικό πρόεδρο της χώρας. Είχαμε και τον κύριο Μπίσλι που μας έλεγε για την ανθρωπιστική κρίση στη χώρα, λέει ο πρόεδρος, μια από τις πιο δραματικές κρίσεις που έχουμε γνωρίσει. Κυρία Λορένσο, καλώς ήρθατε. Με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε την ενημέρωσή σας για την κατάσταση την πολιτική και ανθρωπιστική στη Βενεζουέλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για τη δυνατότητα να σας δώσω μια ενημέρωση. Ε, το πολιτικό αδιέξοδο συνεχίζεται στη Βενεζουέλα. Όπως τα γνωρίζετε, έχει μειωθεί το περιθώριο πολιτικής συνεννόησης και ο αντίκτυπος ανθρωπιστικά και οικονομικά είναι τεράστιος. Διακυβεύεται η ίδια η σταθερότητα της περιοχής. Και παρόλα αυτά βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Θα πω δύο λόγια αρχικώς σχετικά με τον αντίκτυπο στον λαό της Βενεζουέλας. Ξέρετε τους αριθμούς, 10 με 12 εκατομμύρια Βενεζολάνοι έχουν ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια. Σχεδόν 90% του πληθυσμού βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας και με βάση συντηρητικές εκτιμήσεις 6,8 άνθρωποι υποσυτίζονται, 20% του πληθυσμού και πάνω από 50% των παιδιών δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Οι επιπτώσεις, ξέρετε, είναι ότι 5.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν την χώρα και η αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες έχει πλέον μετρήσει 5 εκατομμύρια μετανάστες και πρόσφυγες από τη χώρα και η πραγματική αριθμή μάλλον είναι ακόμα υψηλότερη. Όλα αυτά σε ένα πλαίσιο βαθιών, πολιτικών και συνταγματικών θεσμικών προβλημάτων και δεν έχουμε καμιά ένδειξη να πιστέψουμε ότι αυτοί, αυτές οι ροές εκτοπισμού θα ανασταλούν. Υπάρχει πρόβλημα με την πρόσβαση σε υγειονομικές ε, υπηρεσίες, ε, φάρμακα, τρόφιμα, νερό και προστασία. Για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είπε και ο Ήπατος, ε, εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι παραβιάσεις είναι πολύ σοβαρές Ξέρετε ότι η Βενεζουέλα είναι μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έχει υποχρέωση να τηρεί αυστηρότατα πρότυπα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ακολουθεί τις διαδικασίες που προβλέπει το Συμβούλιο αυτό. Αυτό όμως επιτρέπει από την άλλη μεριά το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση και δραστηριότητα στην Βενεζουέλα. Και παρότι δεν είναι ιδανικά τα πράγματα, είναι αλήθεια ότι βρίσκονται εκεί, είναι το μοναδικό διεθνές ε, σώμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκεται στη Βενεζουέλα και είχε πρόσβαση μέχρι και στις στρατιωτικές φυλακές. Τώρα, όσον αφορά την ε, πολιτική κατάσταση, την παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες. Ξέρουμε, ξέρετε όλοι τα γεγονότα της 5ης Ιανουαρίου και τις προσπάθειες του καθεστώτος να ελέγξει την Εθνοσυνέλευση εκφοβισμός και καταστολή κατά μελών του Συνέλευσης έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, ιδίως ε, με την εκμετάλλευση των κολεκτίβων. Ενώ ο πρόεδρος Γουαϊδό βεβαίως βρίσκεται στη θέση του, αριθμός συμβούλων του αλλά και συγγενείς του έχουν ε, κρατηθεί, ανακριθεί. Δεν φαίνεται να υπάρχει χώρος διαπραγμάτευσης. Παρ' όλα αυτά πρέπει να αποφύγουμε μη αντιστρέψιμες ε, ενέργειες που θα μπορούσαν να ε, εξαλείψουν ε, ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες διαπραγμάτευσης ή εξέβρεσης λύσης. Πρέπει λοιπόν να συγκεντρώσουμε προσπάθειες από διεθνείς φορείς για να αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε παράθυρο ευκαιρίας που θα μας δοθεί μέσω της διενέργειας κοινοβουλευτικών εκλογών του 2006. Σε αυτό περιλαμβάνεται και μια συμφωνία για την, τον ορισμό ε, αξιόπιστης εκλογικής, εκλογική, ε, Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής. Θέλουμε όλοι οι βενεζουελάνικοι φορείς να συμμετάσχουν στην σύσταση, αυτή, στη δημιουργία, την ίδρυση αυτής της ε, Εκλογικής Επιτροπής και αυτό είναι εφικτό η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνεται και σε Βενεζουελάνους ε, εκπροσώπους και σε διεθνείς φορείς. Έχει ε, ε, ενισχύσει τις προσπάθειές της η Ευρωπαϊκή Ένωση στην, <clears throat> στην κατεύθυνση της διενέργειας νόμιμων εκλογών είναι και ο κύριος Ιγκλέσιας στην περιοχή για να συζητήσει διπλωματικούς τρόπους επίλυσης της διαφοράς με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς. Θα πάει και στο Καράκας ο κύριος Ιγλέσιας τις επόμενες εβδομάδες στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών. Βεβαίω η λύση μπορεί να είναι μόνο βενεζουελάνικη, όμως το μέγεθος της κρίσης και οι γεωπολιτικές επιπτώσεις απαιτούν από τη διεθνή κοινότητα να συνεργαστεί με ένα συμπληρωματικό τρόπο ώστε να επιτευχθεί η ειρηνική επάνωδο στη συνταγματική τάξη και την ειρήνη. Φυσικά το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας είναι η ενότητα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αποτύχουν όλα αυτά και το καθεστώς διορίσει η CNA μια τέτοια εκλογική επιτροπή μόνο μονομερός, θα χάσει την ευκαιρία όχι μόνο να, να θεωρηθεί νομιμοποιημένη, αλλά θα απομακρύνει ακόμα περισσότερα την ε, πιθανότητα εκδοχής, εξέβρεσης μάλλον, κοινή ε, λύσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί μέτρα πίεσης ιδίω αν, δεν, αν οι διαπραγματεύσει δεν αποφέρουν καρπούς ή δεν γίνουν κα, καλή τυπίστη. Τα μέτρα μας θα εξαρτηθούν από τις εξελίξει επιτόπου. Να πω και δύο λόγια σχετικά με την αρρωγή που δίνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να δραστηριοποιείται και στον τομέα της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής κρίσης και από το 2018 έχει παράσχει πάνω από 170 εκατομμύρια ευρώ τόσο εντός Βενεζουέλας όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Αν η κρίση έγινε ένα από τα σημαντικότερα σημεία και προτεραιότητες πολιτικής για την περιοχή, παρόλα αυτά ε, δεν έχει τύχει μεγάλης προσοχής στην Ευρώπη. Και η βοήθεια που δίνεται υποχρηματοδοτείται σοβαρά. 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια χρειάζονται στην περιοχή, εκ των οποίων 0% χρηματοδότηση έχει αυτή τη στιγμή εγκριθεί. Η κατάσταση στη χώρα έχει προκαλέσει το μεγαλύτερο εκτοπισμό πληθυσμού στην Αμερική και είναι συγκρίσιμη κατάσταση με εκείνη στη Συρία. Οι Βενεζολάνοι ε, μετανάστες και πρόσφυγες σε άλλες χώρες Λατινικής Αμερικής και της ε, Καραϊβικής έχει αυξηθεί από 123.000 το 2015 σε 4 εκατομμύρια το Δεκέμβριο του 2019. Οι επιχειρικές ε, συνθήκες για τους ανθρωπιστικούς φορείς είναι προβληματικές για πολλούς λόγους οικονομικούς, επιμελητές, ιδίως για διεθνείς και εθνικούς φορείς έχουμε δει μέσα από την, τις ε, ομάδες, την εργασία μάλλον των σημείων επαφής στον ανθρωπιστικό πυλώνα ε, ότι υπάρχει μια σχετική πρόσβαση, ε, βελτίωση στην πρόσβαση. Η συνδιάσκεψη αλληλεγγύης που έγινε στη Βρυξέλλες τον Οκτώβριο αναγνώρισε την επιδεινούμενη κατάσταση στη Βενεζουέλα και αναγνώρισε τις προσπάθειες που κάνουν οι χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες και μετανάστες μέσω του συντονισμού πλαισίου του και έτσι εξαγγέλθηκε και για το πρώτο εξάμεινο του 2020 μία συνδιάσκεψη ε, χρηματοδοτών. Βρισκόμαστε αυτή τη φάση στο, στη διαδικασία εξέβερσης χώρου και χρόνου για τη διεξαγωγή αυτής της ε, συνδιάσκεψης. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, Πρόεδρος. Και τώρα θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων μέχρι τις 5.30, 6 παρατέρτο. Έχουμε δηλαδή, έχουμε χρόνο. Έχω τον κύριο Γκάλα, Μιγιάν Μόν, Τσατσαλιέρος, Τσαβιλόπης, Μάτο, Wallace, Λοιπόν, ο κύριος Γκάλα πρώτα για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ για την ενημέρωση αυτή που είναι απογοητευτική, καταθλιπτική. Ένα καθεστώς τόσο σκληρό όσο αυτό με 5 εκατομμύρια εκτοπισμένους που έχει δημιουργήσει και τις θλιβερές συνθήκες στο εσωτερικό της χώρας μένει να δούμε πώς μπορεί κανείς να υποστηρίξει μια λύση από εκείνους που θα είναι πιο κοντά στα πράγματα. Το πιο σημαντικό πιστεύω είναι να δούμε ότι τα μέτρα που έχουμε αναλάβει θα υλοποιούνται. Τώρα η ερώτησή μου είναι κατά πόσον γνωρίζετε ότι η κυρία που Μαδούρο θεωρεί αντιπρόεδρό του, η κυρία Ροντρίγκε. σταμάτησε για ένα βράδυ στη Μαδρίτη σε διαμετεκόμιση και είχε μια συνάντηση με Ισπανό Υπουργό. Δεν το έχω δίπλο διασταυρώσει, αλλά έγραφαν ότι ξεφορτώθηκαν και 40 βαλίτσες, λέει ο μιλητής. Αυτό δεν θεωρείται ότι είναι κατά παράβαση των μέτρων που είχαμε αναλάβει. Ελπίζω μέσω τέτοιων μονομερών ενεργειών να μην διατεράσετε η ενωμένη μας γραμμή, η ενιαία μας γραμμή και έχουμε και μια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου υπό τη Ρέλεξ για να δει πώς τα διάφορα μέτρα που αναλαμβάνονται στις διάφορες χώρες ε, όπως και στην Ουκρανία και τώρα στη Βενεζουέλα υλοποιούνται. Δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς αποτυπωμένο το θέμα στον τύπο αλλά ε, δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να, να δίνουμε και λανθασμένα μηνύματα ε, στο καθεστώς Μαδούρο και η Ισπανία μάλλον είναι η τελευταία χώρα που πρέπει να κάνει τέτοια πράγματα γιατί τότε θα δοθεί εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, αδιαφορή για το θέμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσαβιλόπες που είναι και συμπρόεδρος της Eurolat. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λορέντσο για τις λεπτομέρειες, για την ενημέρωση της τριβερής κατάστασης που επικρατεί και της πολιτικής που προσπαθούμε να προωθήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση υπό συνθήκες σοβαρότατες, σε αδιέξοδο πολιτικό και σε σοβαρές δυσκολίες ε, να αντιμετωπίσουμε το ακόμη πιο σοβαρό θέμα που είναι το ανθρωπιστικό. Καταστροφικό εσωτερικά και με τεράστιο αντίκτυπο στην περιοχή η οποία έχει μακρύ κατάλογο ελήψεων και προβλημάτων και η ίδια. Ανάγκες δηλαδή του πληθυσμού, όπου στο οποίο ερχόμαστε να προσθέσουμε πλέον εκατοντάδες χιλιάδων, αν όχι εκατομμύρια πρόσφυγες, Βενεζουελάνους. Η Κολομβία, το Εκουαδόρ, το Περού, που ήδη καταβάλουν πολύ σημαντική προσπάθεια ε, υποδοχής μεταναστών και προσφύγων. Ήθελα λοιπόν κάποιες γενικές προατηρήσεις πρώτα να κάνω για τη συζήτηση. Εμείς τακτικά συζητούμε και μάλιστα παθιασμένα. Είναι σοβαρότατη η κατάσταση εκεί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στην προηγούμενη εντολή, θητεία, είχαμε 14 ψηφίσματα. Όμως. Δηλαδή είναι απαραίτητο να συζητούμε το θέμα, αλλά αναρωτιέται κανείς ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά πόσον αφού όλη αυτή η προσοχή που δίνουμε στο ζήτημα χρησιμοποιείται με κάποιον άλλο τρόπο εσωτερικά ή δίνουμε ακόμα περισσότερα μέσα στο καθεστώς, στο καθεστώς μέσω ίσως και άλλων ε, κοινοβουλίων. Εγώ έχω σημαντικές αμφιβολίες για την γραμμή που έχουμε τηρήσει. Είναι σωστό να συζητούμε, καλό είναι να έχουμε ε, να τοποθετούμαστε ανοιχτά, αλλά αν αυτά τα χρησιμοποιούν κάποιοι άλλοι, γιατί ίσως, ε, όπως είπε και ο προηγούμενο συνάδελφο, δεν ξέρω αν μπορούμε δηλαδή ε, ε, επί τέτοια βάση να έχουμε ενιαία γραμμή. Δεν ξέρω αν έχουν συμβληθεί όλα τα κράτη-μέλη προς την, την ενιαία γραμμή που έχουμε ανακοινώσει ότι έχουμε και αναφέρθηκε και ο ύπατος εκπρόσωπος και αναρρύθμιτες φωνές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα είναι πώς θα έχουμε μια ενιαία, κοινή, συμπεφωνημένη θέση που θα υλοποιούν όλοι και που θα είναι χρήσιμη, θα επιφέρει αποτελέσματα για τη Βενεζουέλα. Πρώτον για το ανθρωπιστικό ζήτημα, για την συνδιάσκεψη των δωρητών που ε, διοργανώνεται, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει επιφάνεια στο θέμα αυτό, και δεύτερον, σε μια πολιτική λύση, κλείνω αμέσως πρόεδρε, για το πολιτικό διέξοδο χρειάζεται μια στρατηγική αναγνώριση από όλα τα κράτη-μέλη. Εμείς με επιμέρους κυρώσεις το κάνουμε λίγο πιο κομψά, αλλά κράτη το ε, κάνουν πολύ πιο χονδροειδώς αν θέλετε, για να έχουμε μια προσέγγιση πολιτική ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank you. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Το Renew και το ID και οι πράσινοι δεν ζητούν το λόγο. Η κυρία Φωτίγκα για το ECR. Well, this... Ε, well, this morning... Ε, ε, η κυρία Φωτίγκα σήμερα το πρωί επιμείνατε ότι ο συντονιστής πρέπει να μιλάει πρώτος. Τώρα μου λέτε το αντίθετο από την πολιτική ομάδα, Πρόεδρε, εξαρτάται ποιος θα μιλήσει. Συμφωνήσαμε με τον συνάδελφο ότι θα μιλήσει εκείνος. Δεν είστε απόλυτο συνεπείς όμως, κυρία μου, λέει ο Πρόεδρος. Ε, ναι, Πρόεδρε, είστε πολύ ευγενικός. Δεν χρειάζομαι συμβουλές από πλευρά σας, ε, κυρία Φωτίνκα, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ο κύριος Τέρτς. Εντάξει, έχουμε να κάνουμε με μια καταστροφική κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά από 20 χρόνια τσαβικού σοσιαλισμού ε, όπου τα πράγματα διαρκώς επιδεινώνονται, διαρκώς χειροτερεύουν με τη βοήθεια και της Κούβας προφανώς έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε, έχουμε φτάσει το πιο ε, μισητό καθεστώς που δολοφονεί τους πολίτες του, τους ε, διώχνει από τη χώρα σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο και από τη Συρία και χωρίς να υπάρχει εμφύλιος πόλεμος, ε, ανοιχτός πόλεμος σε πάση περιπτώσει. 30.000 δολοφονίες έχουμε καταγράψει το χρόνο, λέει ο ομιλητής. Είναι όλα αυτά εφιαλτικά. Και υπεύθυνο είναι ένα καθεστώς εγκληματικό καθεστώς, το καθεστώς Μαδούρο, το οποίο δεν έχει καταδικαστεί επαρκώς και δεν έχει υποστεί επαρκείς κυρώσεις. Συνέχισε με τις προκλήσεις του και με τους συμμάχους του. Και τώρα έχουμε με εμφιαλτική κατάσταση. Και ένα πολιτικό κόμμα το οποίο χρηματοδοτείται από τη Βενεζουέλα εισήλθε στην κυβέρνηση στη χώρα μας και κάθεται στο Συμβούλιο Υπουργών. Αυτό είναι ένα πρόβλημα ασφαλείας για την Ευρώπη ολόκληρη, αλλά οπωσδήποτε για την Ισπανία είναι μια τραγωδία. Οι θέσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαιρεμένες γιατί ο κύριος Σάντσεθ αρνήθηκε να υποδεχθεί τον κύριο Γκουαϊντό που τον δέχθηκαν όλες οι χώρες της Ευρώπης και ο κύριος Σάντσεθ δέχθηκε σε μυστική επίσκεψη μία υπουργό που εισήλθε παράνομα στο ευρωπαϊκό έδαφος, που είναι εγκληματίας και κατηγορείται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λαθρεμπόριο ναρκωτικών, λέει ο μιλητής. Έχουμε όλο και περισσότερες αποδείξεις, ενδείξεις ότι έχουμε ένα από τα συγκυβερνώντα κόμματα στην Ισπανία είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη δικτατορία αυτή η οποία πιέζει και το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην Ισπανία διότι και το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει ε, γκρίζες ε, σχέσεις το είχαμε δει και με τον κύριο Θαπατέρο έχουμε μυστικές διασυνδέσεις ε, με το καθεστώς της Βενεζουέλα έχουμε λοιπόν ευρωπαϊκή κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλούμε, υπό εκβιασμό στο χέρι, στο τσεπάκι του κυρίου Μαδόρου. Αυτή είναι η διάγνωσή μου και νομίζω ότι είναι επακριβέστατη, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριος Γουάλλας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Ε, μας ε, δώσετε μια ζωφερή εικόνα της κατάστασης στη Βενεζουέλα. Τα πράγματα όντως είναι προβληματικά εκεί εδώ και αρκετό καιρό. Ήμουνα πέρσι για μια εβδομάδα εκεί και διαπίστωσα ότι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Είπατε ότι η, κατάστα... λύση μπορεί να προέρθει μόνο από το λαό της Βενεζουέλας. Ενώ πιστεύετε ότι υπάρχει και ε, η ανάγκη βοήθειας από τη διεθνή κοινότητα. Εγώ θα έλεγα ότι δεν πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή κοινότητα ήταν πολύ Θα ε, πω ότι ήταν μεγάλο λάθος να αναγνωριστεί ο Γουαϊτό ως πρόεδρος της χώρας. Ε, ενώ ε, διορίστηκε ως αρχηγός της Εθνικής για περίοδο 12 μηνών και μετά αντικαταστάθηκε από κάποιον της δεξιάς, δεν εκλέχθηκε ποτέ και ήταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου ε, να αναγνωριστεί ως ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, εφόσον δεν είχε ποτέ εκλεγεί σε αυτή τη θέση. Ίσως να έχασα αυτά που είπατε, σε αυτά που είπατε, αλλά δεν άκουσα να μιλήσετε για κυρώσεις, ίσως να μην άκουσα εγώ καλά. Αλλά δεδομένων των προβλημάτων στην Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή, ε, δεν είναι αστροφυσική ε, να πει κανείς ότι η μεγαλύτερη επιρροή ε, στην κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα έχει σχέση με τις κυρώσεις της Αμερικής. Οι Αμερικανοί έχουν κάνει τεράστιες προσπάθειες από τον καιρό του Τσάβες τον Ιανουάριο του 1999 να ε, μετατοπίσουν αυτή την κυβέρνηση. Έκαναν, ε, κατάφεραν να υποσκάψουν την τρέχουσα κυβέρνηση με τις κυρώσεις και οι κυρώσεις είναι δρακόντιες. Ε, έχουν πλήξει το λαό, δεν έχουν πλήξει το Μαδούρο, έχουν πλήξει το λαό και έχουν διώξει το λαό από τη χώρα για να πάνε να ζήσουν κάπου αλλού. Δεν νομίζετε εσείς ότι η Ευρώπη θα πρέπει να δει ε, την άρση των κυρώσεων. Δεν νομίζετε ότι θα πρέπει να δουλέψετε με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας για να προσπαθήσετε να επιλύσετε ε, μια πολύ βυσχερή κατάσταση, διότι οτιδήποτε έχει δοκιμαστεί μέχρι στιγμής δεν έχει αποτέλεσμα από ό,τι βλέπω εγώ. Και ξέρω ότι υπάρχουν ε, δικαιολογικά γραφεία που ασχολούνται με ανθρώπινα δικαιώματα που επιμένουν ότι το διεθνές δίκαιο δεν έχει σε αυτή την ε, κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Θα είμαι στο δεύτερο γύρο για το ΕΛΚ ε, να ε, κρατήσουμε δύο λεπτά, δύο ως τρία λεπτά αναομιλητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν από μερικά χρόνια δώσαμε το Ζαχάροφ στην αντιπολίτευση της Βενεζουέλας και ακούμε τώρα αναφορές ότι αυτό δεν τη χάνει σεβασμού, ότι αυτή η αντιπολίτευση ε, ε έχει δυσκολ... πολλές δυσκολίες στη Βενεζουέλα όπου υπάρχουν παραβιάσεις καθημερινά ανθρωπινών δικαιωμάτων. Έχετε εισαγάγει κυρώσεις στην κυβέρνηση. Ποια είναι τα μέτρα που η ΑΕΔ λαμβάνει για την ενημέρωση ε, της κυβέρνησης ότι παραβιάζουν ε, τις κυρώσεις. Ε, ε ναι, η κυρία Σάντσες ήταν στο αεροδρόμιο Μπαράχας και είχε συναντήσεις που δεν πρέπει να είχε. Έχει ενημερωθεί ότι έχει παραβεί τις κυρώσεις και ποια μέτρα μπορείτε εσείς να πάτε για να ενημερώσετε το θέμα αυτό. Λοιπόν, Ευχαριστώ, κύριο Σάντσε eh, eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση που δεν είναι καινούρια. Τα γνωρίζουμε αυτά. Δεν φαίνεται να έχουμε διέξοδο. Πρέπει να εναποθέσουμε όλες μας τις ελπίδες σε αυτές τις εκλογές. Και με αντικειμενικό στόχο αυτήν τη νέα εκλογική επιτροπή όλες αυτές οι ανθρωπιστικές ε, τυχές, ε, το προσφυγικό κτλ. Και η χρήση στην αίθουσα αυτή του ζητήματος Βενεζουέλας, ε, όπως έδειξε περίτρανα ο συνάδελφος Τέρτς, με εσωτερικές μικροκομματικές στοχεύσεις. Μπορεί κάποιοι να χαίρονται να είναι τέτοια πράγματα, αλλά όλα αυτά είναι πολύ θλιβερά που συμβαίνουν εκεί προσπαθούμε με κάθε τρόπο να διατηρήσουμε την ενότητα κριτηρίων και δράσεως. Τώρα, αναφέρεστε εδώ πέρα ε, στην υλοποίηση των κυρώσεων και αυτό αντιστοιχεί στα κράτη-μέλη, ήδη το είπε ο κύριος Μπορέλα. Αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την ε, ε, για το πόσο ειλικρινή είναι η στάση της Α ή της Β κυβέρνησης υπάρχει κατάλληλος χώρος να γίνει αυτό και δεν είναι εδώ. Γιατί τότε αμφισβητείτε την ειλικρίνεια της ανησυχίας για το πρόβλημα της Βενεζουέλας ή τη χρήση του για εσωτερικούς κομματικούς στόχους. Δεν νομίζω ότι μας βοηθάει καθόλου εδώ η τέτοια αναφορά και δεν βοηθάει καθόλου και τη χώρα αυτή όλη αυτή η φαντασιακή τοποθέτηση του κυρίου Τέρτς ότι ο Μαδούρο κάθεται στο Συμβούλιο των Υπουργών της χώρας μας ε, ε, ότι υπάρχουν πρέσβεις που αποστέλλονται μυστικά για να υποστηρίξουν τυραννικές δημοκρατίες, όλα αυτά είναι φαντασιακά. Και ζητώ συγγνώμη και από συναδέλφους άλλων χωρών γιατί ήθελαν σήμερα να συζητήσουν το πρόβλημα της Βενεζουέλας γιατί τους απασχολεί και όχι επειδή θεωρούσαν ότι αυτό είναι ένα καλό παράθυρο ευκαιρίας για να κατηγορήσουμε την σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς από την αρχή προσπαθούμε να αποφύγουμε μια διπλωματική κρίση και ένα διπλωματικό αδιέξοδο σε σχέση με την είσοδο της κυρίας Ροντρίγκε σε ισπανικό εδαφός, την οποία δεν επιτρέψαμε. Σας ευχαριστώ. κυρία Φωτίγκα έχει το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει η κυρία Φωτίγκα. ήταν ο πρόεδρος Μαδούρο και ο προκάτοχός του που οδήγησαν μια χώρα δυνητικό παράδεισο με τεράστιες δυνατότητες πόρων, κλίματος, εργατικού προσωπικού εξειδικευμένου στην καταστροφή, στο μαρασμό σε μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις οπουδήποτε στον πλανήτη. Ήθελα να θυμίσω στους συναδέλφους που μιλούν για διεθνές δίκαιο ότι η διεθνής κοινότητα, λέει η ομιλήτρια, είχε τεράστιες επιφυλάξεις και δώσαμε και το, βραβείο, το βραβείο Ζαχάροφ ε, στην κοινοβουλευτική αντιπολίτευση της Βενεζουέλα υποχρεούμαστε να δείξουμε αλληλεγγύη προς τους συναδέλφους μας, ομολόγους μας που εκπροσωπούν την κοινότητα, την κοινωνία της Βενεζουέλας. Και όπως και η κυρία πρέσβης μας είπε ότι η, η στενή, ο στενός κύκλος, ο οικογενειακός του κυρίου, του κυρίου Γκουαϊντό έχει υποστεί τεράστιες πιέσεις για να μην πω τρομοκρατία. Επομένως, ποιο είναι το επίπεδο στήριξης σήμερα, τώρα, υπέρ του κυρίου Γκουαϊντό. Ποια είναι η παρουσία ξένων φορέων στη Βενεζουέλα. Γνωρίζουμε ότι οι Ρώσοι ήταν εκεί και η παρουσία τους είναι ακόμα εμφανής. Άλλοι υπάρχουν. Να πάμε στους υπόλοιπους ομιλητές, λέει ο Πρόεδρος, από το ΕΛΚ. Ο κύριος Μιαμών, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την εκπρόσωπο της ΙΕΔ για την ενημέρωση την επικαιροποίηση αυτή τη ενημέρωση για τη Βενεζουέλα συμπεριλαμβανομένη τη ανθρωπιστική κατάσταση που είναι πραγματικά λυπηρή. Που προέρχεται από τη διαφθορά τη κυβέρνηση, ε, από το ανελεύθερο αυτό καθεστώς. Ε, δεν χρειαζόμαστε άλλες αιτιάσει, ε, αιτιολογίες. Αυτές είναι. Τώρα, προκειμένου να μπορεί να αξιολογήσει κανείς μια νέα προσπάθεια διαλόγου για τον Μαδούρο ή με τον Μαδούρο, μέχρι στιγμή όλες οι συμμετοχές από πλευράς του ήταν να κερδίσει, για να κερδίσει χρόνο ή για να τα χρησιμοποιήσει εσωτερικά. Θυμίζω ε, Δημοκρατία, Μπαρμπάδο και τα λοιπά, όλες αυτές οι απόπειρε διαμεσολάβησης δεν τηρήθηκαν οι συνταγματικές διατάξεις, φυλακίστηκαν μέλη της οικογένειας του Γκουαϊντό, δηλαδή και τον περασμένο μήνα το κοινοβούλιο αυτό ε, είχε ζητήσει την επέκταση των κυρώσεων για παραβιάσεις κατά συγκεκριμένων προσώπων. Τώρα για την Υπουργό της Βενεζουέλας δεν μας είπε τίποτα η εκπρόσωπος της ΙΕΔ. Ε, τέλος πάντων, ε, ε, δεν ξέρω αν ασχοληθήκατε ακριβώς με, την, με, το, με τη διαμετακόμιση από ισπανικό έδαφος της Υπουργού αυτής της Αντιπροέδρου της Βενεζουέλας, η οποία απαγορεύεται από απόφαση του Συμβουλίου. Η ίδια η διαμετακόμιση, όχι η, προσγείωσή της, η επίσκεψή της. Υπάρχει και ομάδα εργασίας του Συμβουλίου υπό την Ρέλεξ, η οποία ζήτησε ενημέρωση από τις Ισπανικές Αρχές για αυτήν την προφανώς παραβίαση, παράβαση της απόφασης του Συμβουλίου. Η εντολή της Ρέλεξ για τις κυρώσεις συμπεριλαμβάνει και διαβάζω την απόλυτη ενημέρωση σχετικά με όλα τα περιοριστικά μέσα που, έχει λάβει, που έχουν λάβει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομάδα Ρέλεξ ζήτησε πληροφορίες ε, ρωτώ από τις Ισπανικές Αρχές, θα το κάνει. Μίλησε με την ΙΕΔ, μίλησε με την Κροατική Προεδρία, που φαντάζομαι ότι συντονίζει και τη Ρέλεξ. Η ΕΔ θα αναλάβει κάποιο μέτρο προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί ανεξάρτητα από την Επιτροπή υπήρχε και στο Κοινοβούλιο μια συζήτηση. Στο Συμβούλιο πάντως είχαμε σαφείς αποφάσεις. Εν πάση περιπτώσει. Για τις βαλίτσες ήδη, ήδη είπε ο συνάδελφος, δεν, μπορώ, δεν έχω άλλο χρόνο να ασχοληθώ, αλλά θα ήθελα να καταλάβω. Η διαμετακόμιση αυτή έλαβε χώρα, θα λάβετε μέτρα. Ενημερωτικά. Ευχαριστώ κύριο Σαρθαλέχος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πριν από λίγες ημέρες, η αντιπρόεδρος της Ισπανικής κυβέρνησης σε ευνηδιαστική ανακοίνωση είπε ότι η Βενεζουέλα δεν ενδιαφέρει κανέναν. Και το λέω, το παραθέτω. Εμείς έχουμε διαφορετική άποψη ελαφρώς. Εμείς θεωρούμε ότι η Βενεζουέλα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι προτεραιότητα και βεβαίως και μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να υποστηρίξουμε τη δημοκρατία στη χώρα αυτή και μας ενδιαφέρει λόγω της τραγικής αυτής ανθρωπιστικής κρίσης της οποία διέρχεται η χώρα αυτή. Το θέμα των κυρώσεων είναι σίγουρο ότι η χειρότερη κύρωση και που πρέπει να αρθεί είναι αυτή που επιβαρύνει τους κατοίκους της Βενεζουέλας που καταπιέζονται από ένα απολυταρχικό καθεστώς. Καταπιέζονται πολιτικά και οικονομικά. Και όπως θα γνωρίζετε και εσείς, αναφερθήκαμε στην παραβίαση από πλευράς αντιπροέδρου της Βενεζουέλας, όπου την υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο Μπαράχας υψηλό, υψηλό βαθμός τέλεχος της Ισπανικής κυβερνήσεως. Αυτό το θέμα, παρότι παρουσιάζεται ως κομματική αντιπαράθεση, δεν είναι. Εχθές εχθές δικαστής στη Μαδρίτη ζητήθηκε ε, διέταξε να, να παραδώσουν τις μαγνητοσκοπήσεις των ε, καμερών ασφαλείας του αεροδρομίου για να δει κατά πόσον υπήρχαν ενδείξεις ποινικά κολάσιμης πράξεως κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής. Δηλαδή τα πράγματα επιδεινώνονται μέρα με τη μέρα. Έναντι λοιπόν αυτή τη κατάσταση που επιδεινώνεται καθημερινά φαίνεται ότι να είναι ασυγχώρητο η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των μηχανισμών αναφέρθηκατε ήδη στην ηρέλεξη και στο σύστημα κυρώσεων αν μη τι άλλο πρέπει να ζητάει ενημέρωση, πληροφορίε. Εμεί είμαστε απόλυτο υπέρ τη κοινή γραμμή και θέση για τη Βενεζουέλα αλλά αυτή η κοινή γραμμή και θέση προϋποθέτει την απόλυτη και χωρίς αμφιβολίες αναγνώριση του ως μεταβατικού προέδρου του κυρίου Γκουαϊντό και την επιβολή του συστήματος κυρώσεων. Η ισπανική κυβέρνηση και στα δύο αυτά λυπούμε αλλά δεν συμμορφούνται. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λόπες που γνωρίζει την κατάσταση και τη χώρα αυτή εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Έχοντας ακούσει τις τοποθετήσεις σήμερα, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αναγκαιότητα να εξηγήσουμε γιατί είναι ενδιαφέρουσα σημαντική η Βενεζουέλα για το Ευρωπαϊκό αυτό κοινοβούλιο. Ίσως ε, είναι χρήσιμο να σας εξηγήσουμε γιατί είναι μεταβατικός πρόεδρος ως πρόεδρος της ε, Εθνικής Συνέλευσης ο κύριος Γκουαϊντό μετά την εκλογή του επανεξελέγει. Επανεξελέγει ο κύριος Γκουαϊντό. Μετά την απόπερα του καθεστώτος να κλείσει τη Βουλή. Όσοι ανησυχείτε για τις κυρώσεις, ότι αυτό θα μπορούσε να είναι τιμωρία για τους πολίτες και όχι το καθεστώς, θυμίζω ότι όταν το καθεστώς του Τσάβες ή του Μαδούρο όλα τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή, τα 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τα χρησιμοποιούσαν, σήμερα είναι περί 100.000. Αυτό είναι η πηγή του προβλήματος. Όπως και η εκμετάλλευση των ε, ε ορυχείων χρυσού και, και η ο αναγκαστικός εκτοπισμός των ε, Ινδιάνων Ιθαγενών. όλα αυτά ήταν ο μόνος τρόπος που βρήκε το καθεστώς για να κερδίσει χρόνο που ήταν η απόλυτη προδοσία προς τον λαό της Βενεζουέλας. Δεν πρόκειται να καταλήξετε σε κανένα αποτέλεσμα με οποιαδήποτε προσπάθεια διαλόγου γιατί δεν τηρεί τις υποσχέσεις του το καθεστώς. Παρά μόνο με τις κυρώσεις οι οποίες θα πρέπει να επιβληθούν αυστηρά και χωρίς να εξαιρείται κανένα κράτος μέλος. Μόνο με τις κυρώσεις θα μπορέσετε να επιτύχετε, να ασκήσετε πίεση στον κύριο Μαδούρο και να αφήσει επιτέλους την εξουσία, λέει ο Μιλτής. Ευχαριστώ. Μάτο. de, de Venezuela, yo pienso... εγώ σκέφτομαι τις Κανέριες νήσους όταν μιλούμε για τη Βενεζουέλα, διότι υπάρχουν χιλιάδες κάτοικοι από εκεί που έχουν επιστρέψει. Είναι πολλά χρόνια που μιλούμε για τη Βενεζουέλα. Ότι βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, ότι υποφέρει ο λαός. Και υπάρχει το εξής παράδοξο. Η κυρία Ροντρίγκεφ ε, έχει απαγόρευση εισόδου στο έδαφος Σέγγεν. παρόλα όλα αυτά εισέρχεται στο ισπανικό έδαφος, πάει στο αεροδρόμιο, συναντάται με υπουργό της Ισπανικής κυβέρνησης. Παραλλήλως, πολύ πρόσφατα, αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χωρίς να έχει κανένα περιορισμό μετακίνησης, εφτάνει στο αεροδρόμιο της Βενεζουέλα, μας κλείνουν σε μια μικρή αίθουσα και μετά μας αποβάλλουν. Μας απομακρύνουν από τη χώρα. Δεν μας επιτρέπουν την είσοδο. Αυτά είναι παράδοξα, δεν είναι. Τώρα, ο κύριος Λόπεθ το είπε πολύ σωστά η λύση δεν είναι διαπραγμάτευση ή η επιτροπη ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά είναι παγίδες, απατηλά. Δεν θα οδηγήσουν στην δημιουργία συνθήκων ελεύθερων εκλογών στη Βενεζουέλα. Γιατί η παράνομη κυβέρνηση της ε, Βενεζουέλας δεν θα το επιτρέψει αυτό. Υπάρχει δέσμευση. Βεβαίως και υπάρχει. Υπάρχει η δέσμευση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το οποίο επικαλείται ο Μαδούρο ως μυστικό. Την παράνομη συνάντηση. Και τι έγινε με αυτές τις 40 περίεργες βαλίτσες που ξεφορτώθηκαν. Θα πρέπει να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί υπάρχει ο ύπατος ε, ε, εκπρόσωπος, υπάρχει η αντιπρόεδρος, υπάρχουν όλα αυτά τα αντιφατικά μηνύματα και υπάρχει και η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως το κάνει σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις, να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να τηρούν τα συμπεφωνηθέντα στο Συμβούλιο. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και νομική δέσμευση. Διότι διακυβεύεται και η αξιοπιστία και αυτού εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Πάολο Ραντζέλ. Στέρνε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν ήδη στην ανθρωπιστική κατάσταση. Εγώ θέλω να θέσω ένα άλλο, πολύ συγκεκριμένο όμως ερώτημα. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αποφάσισε αυτήν την εβδομάδα να απαγορεύσει τις πτήσεις της εταιρείας TAP, της πορτογαλικής εταιρείας, με πρόφαση ότι δεν εξασφαλίζονται οι κανόνες ασφαλείας, γιατί υποτίθεται ότι υπήρξε περίπτωση όπου με πτήση της συγκεκριμένης εταιρείας μεταφέρθηκαν εκρηκτικές ύλες από τον θείο του μεταβατικού προέδρου ε, ο οποίος κατηγορείται ότι έκανε κάτι τέτοιο για να τα μεταφέρει στο Καράκας. Είναι πραγματικά διανόητο το να εκτοξεύονται τέτοιες ε, κατηγορίες και να μην μπορεί να βρεθεί μια λύση. Επαναλαμβάνω ότι ακόμη δεν επιτρέπεται στις ε, στα αεροσκάφη της ΤΑΠ να προσγειωθούν στο Καράκας, κάτι που μου φαίνεται τελείως ακατανόητο. Απαιτούμε την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Πορτογαλία. Γιατί η μεγαλύτερη εθνική μειονότητα που ζει στη Βενεζουέλα είναι Πορτογάλοι ή τέλος πάντων απόγονοι Πορτογάλων οι οποίοι επίσης είναι εξαιρετικά ανήσυχοι λόγω αυτής της κατάστασης. Γιατί είναι σαν να λέει κανείς ότι το, η Πορτογαλία συμμετέχει σε κάποια κρυφή συνωμοσία εναντίον του Μαδούρο. Δεν γίνεται να τα δεχτούμε αυτά. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει συγκεκριμένη θέση. Είναι μια ε, απόφαση αυτή των ε, αρχών της Βενεζουέλας που αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορά την Πορτογαλία, τη συγκεκριμένη εταιρεία και ιδίως όλους εκείνους που πλήττονται από την κρίση. Υπάρχει και ισπανική μειονότητα και ιταλική μειονότητα στη Βενεζουέλα. Όλοι αυτοί πλήττονται από την ε, κρίση και από το καθεστώς. Και τέλος ο κύριος Ταγιάννη, εκ μέρους της ε, διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το κοινοβούλιο αυτό ήταν ο πρώτος διεθνής φορέας και ο πρώτος φορέας στην Ευρώπη που αναγνώρισε ως μεταβατικό ηγέτη τον κύριο Γκουαϊντό. Εμείς υπερασπιστήκαμε πάντοτε τη δημοκρατία, δώσαμε το βραβείο Ζαχάροφ στην αντιπολίτευση της Βενεζουέλα, αλλά δεν είδαμε αντίστοιχη θαραλέα κίνηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσεως. Πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις ε, σε αυτούς που εξακολουθούν να περιορίζουν την ελευθερία του λαού της Βενεζουέλα. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να γίνει κατανοητό ότι πρέπει να πάμε προς μια εξομάλυνση, έναν εκδημοκρατισμό. Υπάρχει και το άλλο θέμα της κυκλοφορίας του ευρώ στη Βενεζουέλα. Υπάρχει η κεντρική τράπεζα που προωθεί την κυκλοφορία χρυσού, ίσως σε ευρώ, ίσως και με τη συνεργασία κάποιων ε, κρίσεων από την Τουρκία για να κάνουν δεν ξέρω και εγώ τι. Εγώ 28 Οκτωβρίου ζήτησα από τον ύπατο εκπρόσωπο ενημέρωση σχετικά με αυτό και ακόμα περιμένω. Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, τέσσερις μήνες περάσανε, ούτε κουβέντα δεν ακούστηκε από τον ύπατο εκπρόσωπο. Δεν μπορεί να προσποιούμαστε ότι δεν ξέρουμε, δεν είδαμε δεν ακούσαμε έναντι και εν πάση περιπτώσει εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θεσμικών εκπροσώπων. Δηλαδή, υπάρχει υποχρέωση και υπό τη συνθήκη να απαντάτε όταν σας γίνονται ερωτήσεις. Τι συμβαίνει με τα χρήματα που έχουν καταλήξει στη Βενεζουέλα, τι τα κάνουν αυτά τα φιλεράκια του Μαδούρο. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές. Ακούσαμε όμως πολλούς συναδέλφους, οπότε θα έχετε την ευκαιρία τώρα να απαντήσετε σε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις. Έχουμε άλλα 15 λεπτά. 6 παρα 5 πρέπει οπωσδήποτε να κλείσουμε. Ευχαριστώ. Έχουμε καταγράψει βεβαίως όλες τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν. και για την ε, επίσκεψη της Τέλση Ροδρίγες και την εικαζόμενη παραβίαση της επιβολής κυρώσεων. Ξέρετε ότι και εγώ θα δώσω περίπου την ίδια απάντηση που έδωσε ο υπάτος εκπρόσωπος στην Ολομέλεια ότι, και θα υπενθυμίσω ότι η τήρηση των περιοριστικών μέτρων που έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Όσον αφορά την Ρέλεξ, Θα έλεγα ότι σε περίπτωση ταξιδιωτικών απαγορεύσεων αυτά παίρνουν, αυτές παίρνουν τη μορφή απόφασης του Συμβουλίου που είναι δεσμευτική για τα κράτη-μέλη. Όμως, αντίθεση με άλλα περιοριστικά μέτρα, μια ταξιδιωτική απαγόρευση δεν περιλαμβάνεται σε κανονισμό του Συμβουλίου που μπορεί να επιβάλλει άμεσα ε, απαγορεύσεις όσον αφορά την είσοδο ατόμων στην Ένωση. Αποσία λοιπόν κανονισμού, η Κομισιόν δεν μπορεί να ελέγξει ούτε να ξεκινήσει τη διαδικασία επί παραβάση. Αυτή είναι η απάντηση που μπορώ να σας δώσω. Ξέρετε ότι έχουμε περιοριστικά μέτρα. Η Ντέλση Ροντρίγε βεβαίω υπόκειται σε τέτοιο περιοριστικό μέτρο, όμω η εφαρμογή αυτού του περιοριστικού μέτρου εναπόκειται στα κράτη-μέλη και μόνο. Νομίζω ότι απάντησα με αυτή τη μία απάντηση που έδωσα σε διάφορες ερωτήσεις που ακούστηκαν. Κύριε Γόλας, για τις κυρώσεις. Οι δύο σημαντικές παρατηρήσεις που θέλω να κάνω είναι ότι οι κυρώσεις που έχουμε επιβάλει ως Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν, είναι εξατομικευμένες κυρώσεις. Έχουμε 25 μέλη του καθεστώτος, αν θέλετε, Μαδούρο, που συνδέονται με σοβαρότατο τρόπο με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτές οι κυρώσεις δεν έχουν καμία απολύτως επίπτωση στον λαό της Βενεζουέλας. Εμείς, σε αντίθεση με Τσίπα, δεν θεωρούμε ότι οι κυρώσεις είναι το μοναδικό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας. Είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Θα παρατηρούσα όμως ότι αν δείτε τα στοιχεία και τις οικονομικές μελέτες, η, κατάσταση, η οικονομική κατάσταση της ε, Βενεζουέλας ήταν πολύ κακή ήδη και πριν από την επιβολή καιρώσεων. Βεβαίω, κάποιες από τις κυρώσει των ΙΠΑ σε εταιρείε και σε συγκεκριμένες δραστηριότητε στην ε, Βενεζουέλα σίγουρα θα επέτειναν και θα όξυναν την ε, δυσκολία, τις δυσκολίες, τις αντικσότητες που αντιμετωπίζει ο λαός της Βενεζουέλας. Όσον αφορά το επίπεδο στήριξης ε, στον Χουάν Γουαϊδό, είναι ε, ενδιαφέρον θα έλεγα αυτό το ερώτημα. Τα στοιχεία που έχουμε λάβει τα τον τελευταίο καιρό ποικίλουν πριν από ένα χρόνο ο Γουάν Γαϊδό είχε ποσοστό έγκρισης, δημοτικότητας αν θέλετε, ε, μεταξύ του βενεζουλάνικου λαού γύρω στο 60%. Ήταν ισχυρός. Όμως το γεγονός ότι δεν κατάφερε να επιβάλλει ή να επιφέρει, να επιφέρει τις αλλαγές που υποσχέθηκε σε έναν λαό που βρίσκεται αντιμέτωπος με τον καθημερινό αγώνα επιβίωσης η δημοτικότητά του έχει καταρρεύσει. Από 20% ακούμε έως 40% ποσοστό έγκρισης. Βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν ανέρχονται τα ποσοστά δημοτικότητάς του σε εκείνα που είχε ο ίδιος πριν από ένα χρόνο. Υπάρχει λοιπόν μια πτώση όσον αφορά στην υποστήριξη Τη ε, αντιπολίτευσης ακριβώς γιατί δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί η αντιπολίτευση στις ε, εξαγγελίες της. Όσον αφορά την παρουσία εξωτερικών φορέων παραγόντων ε, πράγματι υπάρχουν και τους γνωρίζουμε. Η Ρωσία και ο Πρωθυπουργός Λαυρόφ έχουν επισκεφθεί πρόσφατα την Βενεζουέλα. Ξέρουμε ότι εμπλέκονται βεβαίως και προβαίνουν και επιδίδονται και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Βενεζουέλα. Οι χθεσινές αμερικανικές κυρώσεις εναντίον του Ρόσνιευ βεβαίως εντάσσονται στην ευρύτερη αυτή εικόνα. Η δική μας προσέγγιση είναι ότι προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι οικονομικά και πολιτικά στα, ε, της Βενεζουέλας και εκεί πράγματι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα όταν η συνολική συζήτηση δεν έχει ένα συγκεκριμένο στόχο, μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Εμείς λοιπόν η στάση μας είναι ότι θέλουμε να παροτρύνουμε τη διεθνή κοινότητα, αν όχι να έχει μια ενιαία στάση, να αποστέλει τουλάχιστον ένα συνεπές και συνεκτικό ε, μήνυμα όσον αφορά την ανάγκη να υπάρξει ε, μια, να σημειωθεί πρόοδος μέσω του οχήματος της διαβούλευσης και της διαπραγμάτευσης. Και τέλος, ξέρουμε ότι έχει επιβληθεί αυτός ο περιοριστικός όρος στην ΤΑΠ για 90 ημέρες. Νομίζουμε ότι αυτό είναι μια απόφαση που ελήφθη χωρίς τη δέωσα επιμέλεια, που νομίζουμε ότι είναι αντικείμενο ε, πολιτικής εκμετάλλευσης. Νομίζω ότι σε καμία περίπτωση η αναστολή αυτή των πτήσεων της ΤΑΠ ε, μπορεί να γίνει αποδεκτή. Όσον αφορά ε, την επιστολή που στείλατε, κύριε Τέρης, είναι πολύ δύσκολο να απαντήσουμε. Γιατί παρά το γεγονός ότι κυκλοφορούν πάρα πολλές φήμες στην Βενεζουέλα, για χρυσό, το ανέφερε και ο Χουάν Γουαϊδό, για 40 βαλίτσες χρυσού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβεβαιωθούν αυτές οι φήμες. Ε, δεν έχουμε κανένα στοιχείο αυτή τη στιγμή για να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο. Και αν δεν έχει στοιχεία προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξεις σε ασφαλή συμπεράσματα ή να με μετουσιώσεις τις φήμες αυτές σε πραγματικά στοιχεία. Αλλά εργαζόμαστε και επ' αυτών των θεμάτων. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Υπάρχουν ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν. Ο κύριος Μάτο. Τι γίνεται με αυτές τις βαλίτσες ε, της Υπουργού, που, που βρίσκονται και, τι, και τι, τι βρισκόταν μέσα σε αυτή, ποιο ήταν το περιεχόμενο αυτών των βαλίτσων, ε, δεν έχετε στοιχεία, απαντάει ε, η εκπρόσωπο τη ΕΕΔ. Όχι μόνο δεν έχουμε στοιχεία, δεν ξέραμε καν ότι υπάρχουν. Έχουμε άλλα 9 λεπτά, λέει ο πρόεδρο, οπότε μπορώ να δώσω το λόγο στον ε, κύριο Μάτο, τον κύριο Μιλαμόν και τον κύριο Ράνχελ. Όχι, εγώ δεν θα πω για τι βαλίτσε. Απλώ, ε, όπω αναφερθήκατε και εσεί για την επιτήρηση και τον έλεγχο ότι πρέπει όλα αυτά να είναι αποτελεσματικά και εξαρτάται από το κράτη-μέλη. Οπότε, ερώτηση. Έναντι κατάφορης παραβίασης από πλευρά κράτου μέλου, τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να κάνουν τίποτα σε μια τέτοια περίπτωση. Τίποτα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μιαμών. Αν σας κατάλαβα καλά, πρόεδρε, μάλλον κύρια μου, το, η ομάδα Ρέλεξ δεν έχει αρμοδιότητα, αν σας καταλαβα καλά. Ο κύριος Μπορέλ στην Ολομέλεια δεν αναφέρθηκε στη Ρέλεξ, αλλά είπε και παραθέτω η ΕΔ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή όπου έχει αρμοδιότητα θα είναι σε άμεση επαφή με τα κράτη-μέλη σε σχέση με υποτιθέμενες παραβιάσεις ώστε οι κυρώσεις να εφαρμόζονται ομοιογενέως όλα τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, ο κύριος Μπορέλ ε, θεωρεί ότι η ε, ΕΔ κατά κάποιον τρόπο έχει μια αρμοδιότητα αν μη τι άλλο παρακολούθησης επιτήρησης. Εσείς μας είπατε ότι η ομάδα Ρέλεξ δεν έχει αρμοδιότητα. Ούτε η ΕΔ έχει. Γιατί μόλις σας διάβασα τη δήλωση του κυρίου Μπορέλ στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα και επομένως υπάρχει μια αρμοδιότητα επιτήρησης από πλευράς η Τώρα δεν ξέρω επί τη βάση κανονισμού ή απόφαση ή τι, αλλά υπάρχει μια αρμοδιότητα. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπε και ο κύριος Μάτο. Δεν υπάρχει κανένα μέσον επιβεβαίωσης, εξακρίβωσης, επιτήρησης και δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα έναντι τέτοια ε, εμφανούς παραβίασης. Σας ευχαριστώ κύριος ε, Ραντζέλ ε, και πάλι. Ε, πρώτα απ' όλα, Πρόεδρε, να ζητήσω συγγνώμη γιατί χρειάστηκε να βγω για λίγα λεπτά ε, και να πάω στην Αύκο όπου ήμουν με τον Πρόεδρο Ταγιάννη. Για να ζητήσω και από αυτού συγγνώμη δηλαδή. Τέλος πάντων, ναι. Ε, ε, καταλαβαίνω ότι είπατε με σαφήνεια ότι η συμπεριφορά αυτή, η στάση αυτή είναι απαράδεκτη. Τώρα εγώ αυτό που θα ήθελα να καταλάβω είναι αυτό δεν πρέπει να καταστεί δημόσιο ότι είναι δηλαδή απαράδεκτη. Δεν θα έπρεπε να έχουμε μια δήλωση, επίσημη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εν πάση περιπτώσει του υπάτου εκπροσώπου που να καταδικάζει επισήμως την στάση του καθεστώτος Μαδούρο σε αυτήν την περίπτωση. Δηλαδή Καλό είναι που μας βεβαιώνετε με τα λόγια σας, αλλά καθότι εδώ μιλούμε για μια δημόσια δήλωση από το γραφείο του Μαδούρο, πρέπει να έχουμε και μια επίσημη δήλωση από Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι έτσι. Εφόσον δεν ζητάει κανένα άλλο ε, το λόγο, ένα τελευταίο γύρο τοποθέτησε από εσάς. Για να απαντήσω και στις δύο ερωτήσει ε, του κ. Μάτος και του κ. Μιλάν. Ο ύπατος εκπρόσωπος ε, δεν έχει τη δυνατότητα να διεξαγάγει έρευνες στο θέμα παραβιάσεων κυρώσεων. Όμως είναι αρμόδιος για να διασφαλίζει την συνέπεια της ε, χρήσης κοινής πολιτικής ασφαλείας και εκεί μπορεί να εγείρει θέματα που απασχολούν τα κράτη-μέλη ή το Συμβούλιο. Αυτό συνάδει και με αυτό που ελέγχθηκε και στην Ολομέλεια από την είπα εκπρόσωπο. Τώρα, στο θέμα του ΤΑΠ, ναι, εναπόκειται στον είπα εκπρόσωπο να αποφασίσει για δηλώσεις και θα μεταφέρω τις ανησυχίες σας. Σας ευχαριστώ. we can Μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε αυτό το θέμα και εδώ κυρίως και τη λήξη των εργασιών της σημερινής συνόδου. Αύριο θα συνεχίσουμε στις 9 η ώρα και ο Βίτολ Βασικόφσκι θα προεδρεύει την αυριανή σύνοδο. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους που θα πάνε στην Τουρκία την ερχόμενη εβδομάδα να παραμείνουν εδώ, διότι θα ξεκινήσουμε με την προπαρασκευαστική συνάντηση για την επίσκεψη αυτή.